Οι αρμόδιες ε, αρχέ τη Πορτογαλίας έχουν <clears throat> ενημερώσει ότι ο κ. Ζωάου Νούνο Καλάντου Μέντε θα αντικαταστήσει την κυρία Κριστίνα Ζούπερ από την 31η Ιανουαρίου 2016. Το Κοινοβούλιο καταγράφει την ε, ε, τον, την εκλογή του κυρίου Πιμέντα Λόμπες. Τον καλωσορίζουμε και υπενθυμίζω ότι όσο δεν έχει γίνει ο έλεγχο τη εντολή του, απολαμβάνει το πλήρων δικαιωμάτων του ω βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια και στα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Ζίπελ θέλει να λάβει το λόγο για την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένε δηλώσει που έλαβαν χώρα στην Γερμανία και να σας ρωτήσω αν έχετε